The uh, next item on the agenda is the... Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προ τον Βουλή και την Επιτροπή για την επανεκτάση πρωτοβουλία σχετικά με τις ΜΜΕ, Small Business Act. Πρώτο μελίδι έχουμε τον κύριο Μπέντσεν. Για δύο λεπτά. Ως εισηγητή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η οικονομική κρίση είχε επίδραση ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε νέους περιορισμούς που εισάγονται με την οδηγία για τα κεφάλαια. Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να παραγάγουν κεφάλαιο και, και ω εκ τούτου την ανάπτυξη που τόσο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να απευθύνουμε λοιπόν ένα σαφέ μήνυμα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι αποφάσει που απαιτούνται πρέπει να ληφθούν τώρα προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπόθηκε ότι η πολιτική δεν θα πρέπει να είναι ε, πρόεδροι επιχειρήσεων, διοικητικών συμβουλών επιχειρήσεων. Θα έπρεπε όμως να μπορούν να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρούν, να αναπτύσσονται, να ενισχύονται. Αντί λοιπόν να κάνουμε διδάγματα για το πώς θα πρέπει να είναι θα πρέπει να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις αυτές, τις μικρές ιδιαίτερα, στην ε, εδραίωσή τους, στην πρόσβαση στην αγορά, στις συνθήκες ε, λειτουργίες ε, τους, στη συμμετοχή τους στους δημόσιους διαγωνισμούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα εν να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει να περιοριστεί το, ε, ο, δημισ... ο γραφειοκρατικός φόρτος για τις μικρές επιχειρήσεις. Επί παραδείγματι, υπάρχει σύστημα πολλαπλών ε, κοινοποίησεων. Δεν θα μπορούσε να γίνει μόνο το μία φορά η κοινοποίηση και να μην ε, έχουμε τόσο, πολλά, ε, τόσο πολλές διαδικασίες. Αυτό δεν θα επέλυε πολλά προβλήματα. Πολλές φορές τα μέτρα που εισάγουμε στην Ευρώπη, αντί να πλουστεύουν την κατάσταση, την επιδεινώνουν την περιπλέκουν και δυσκολεύουν τα πράγματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν από εδώ και μπρο να φροντίζουμε κάθε τι, κάθε τι που αποφασίζουμε, κάθε νομοθέτημα να μην ενισχύει το φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χερτσόκ. Eh, κύριε Επίτροπε, ρίχνω μια ματιά στο θεωρείο και βλέπω επί, ότι έχουμε επισκέπτες από την ε, Ουγγαρία. Για πέστε μας. Αυτή η πρωτοβουλία σε τι αποσκοπεί. Στην μεταρρύθμιση της ισχυούς νομοθεσίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν 39 διαφορετικά σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είναι σημαντική και η εφαρμογή της νομοθεσίας. Κάποιες χώρες φροντίζουν περισσότερο από άλλες για την υλοποίηση αυτών των μέτρων. Ας πούμε χρειάζεται μια ενιαία βάση δεδομένων για να ξέρουμε πού πάει καλά η υπόθεση και πού όχι. Δεν θέλουμε βεβαίω να παραβιάζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όμως θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να έχουμε δημιουργία θέσεων εργασίας. Θα πρέπει επομένω να πριτανεύσει πνεύμα συνεργασία. Θα πρέπει επίση να μπορούν οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση σε εύκολη χρηματοδότηση. Επίσης να είναι εύκολη η, ε, το να ανοίγει κανείς μια τέτοια επιχείρηση Είπαμε ότι πάμε καλά μέχρι, μέχρι τώρα σε κάποιους τομείς αλλά όχι σε όλους. Είναι πολύ σημαντικό επομένως να δούμε πώς θα υπάρχει η απαραίτητη υποδομή ούτως ώστε να βοηθήσουμε τις ε, επιχειρήσεις αυτές να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρήσεων για να δοθεί μια συνέχεια στο πρόγραμμα Έρασμο ούτω ώστε να βοηθηθούν οι νέοι επιχειρηματίες. Έχουμε 20 εκατομμύρια τέτοιες επιχειρήσεις, πολλές από αυτές απασχολούν έναν ή δύο εργαζομένους. νομίζω ότι θα, αν τι βοηθήσουμε θα βοηθήσουμε την αγορά εργασίας. Επομένως, αυτοί που δουλεύουν στις ΜΜΕ θα πρέπει να έχουν καλύτερη κατάρτιση, καλύτερες δεξιότητες. Αυτό θα βοηθήσει και το πρόγραμμα της πράσινης οικονομίας και επίσης ε, θα πρέπει να ε, βοηθήσουμε να περάσει η ψηφιακή τεχνολογία και στις ΜΜΕ. Ναι, όντω θα πρέπει να καλωσορίσουμε και από αυτή τη θέση του επισκέπτε μα που κάνουν τόσο δρόμο να έρθουν να μας δουν από την Ουγγαρία. Κύριε Χολ. Thank Πρόεδρε, αυτή η πρωτοβουλία ήταν ε, πάρα πολύ καλοδεχούμενοι από τις ΜΜΕ εδώ και μία διετία, άρα είναι σημαντικό. Τώρα θα τους δείξουμε ότι αυτό δεν ήταν μόνο ασκήσεις επί χάρτο. Όσον αφορά τώρα τις διοικητικές υποχρεώσεις, ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι ε, μια ε, επιτυχία που χωρίς συνέχεια θα πρέπει να δοθεί συνέχεια στο θέμα. Ακριβώς οι πιο μικρές αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί το να έχει κάποια επιχείρηση 250 εργαζόμενους, εντάξει, έχει εξειδικευμένους. Όμως, για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ένα-δύο εργαζομένους τότε, η γραφειοκρατία είναι εμπόδιο και έχουμε και πάρα πολλέ. Το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουν κάτω από 10 εργαζομένου επομένω θα πρέπει αυτέ οι πιο μικρέ επιχειρήσει να αντιμετωπιστούν ω οικογένειε. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να εξεταστεί το πώ είναι δυνατόν να βοηθήσουμε αυτέ τι ε, επιχειρήσει και να είναι και πιο ενεργειακά αποτελεσματικέ, γιατί το θέμα τη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να, μόλι πριν το Πάσχα, διάφοροι βουλευτέ τη ε, Ήτρε πήγαν στην ε, Καλιφόρνια να δουν εκεί πέρα στην Silicon Valley τι επενδύσεις γίνονται και είδανε ότι επιχειρηματικά κεφάλαια venture capital κινούνται πολύ πιο εύκολα από ό,τι στην Ευρώπη. Και βέβαια ήταν πολύ πιο ρηψοκίνδυνοι από του Ευρωπαίου. Αυτοί λοιπόν που επενδύουν σε επιχειρήσει λένε ότι 9 στι 10 που δεν τα πάνε καλά, αλλά η δέκατη που θα τα πάει καλά θα αντισταθμίσει τη ζημιά από τι πρώτε 9. Έτσι θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις ε, μείωσες στην Ευρώπη και να μην θεωρούμε ότι είναι ανάθεμα η αποτυχία. Απλά να θεωρείται ένα, μια φάση με ένα σκαλί για να φτάσει κανείς στην επιτυχία. Τσίτσεστερ. Πρώτα ευχαριστώ. Εδώ έχουμε ένα τρομερό παράδοξο στην πολιτική που ασκούμε στην Ένωση για τις ΜΜΕ. Ότι μία μεριά ομόφωνα συμφωνούμε ότι είναι σημαντικές για αγορά εργασίας, οικονομία, καινοτομία, ευελιξία και όσον αφορά το πόσο συμμετέχουν στην οικονομία μας. Και όμως, όταν έχει όλα αυτά να υλοποιηθούν, τότε δεν γίνεται το ίδιο. Η μεγάλη πρόκληση που αυτό το ψήφισμα εντοπίζει είναι το πώς όλα αυτά τα θετικά λόγια θα γίνουν χρήσιμες πράξεις. Χωρίς να διασπαθίζουμε χρήματα, τα οποία χρήματα τόσο σπανίζουν στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Από την άλλη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι αυτές οι καλές προθέσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από μια πολυνομία προστασία περιβάλλοντο και, και, και, διάφορα ωραία πράγματα. Αλλά τελικά έτσι βαραίνουμε αυτέ τι εταιρείε. Το διοικητικό άχθο, α πούμε, είναι τόσο μεγάλο. Θα πρέπει επομένω να τι ξαλαφρώσουμε. Αυτό το ψήφισμα έχει πολλέ θετικέ προτάσει. Ιδίω η πρόταση αυτή που λέει ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική είναι και στη χώρα μου. Οπότε δηλαδή θα, πρέπει, θα μπορούν, να μπορούν οι εθνικές αρχές να προσθέτουν νομοθετήματα ή σε αυτά τα οποία α, θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. οποια αυτή η γραφειοκρατία να συρρυκνωθεί. Όμως, το πιο σωστό που να κάνουμε για να βοηθήσουμε τις είναι να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ε, πληροφόρηση και στην χρηματοδότηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Τσίσεστερ και δίνω το λόγο πρώτα στον κύριο Μπουτικόφερ. Yeah. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν τυχαίνει κάθε μέρα στο Κοινοβούλιο να απευθύνουν έξι, ε, βουλευτές από έξι διαφορετικές πολιτικές ομάδες ερώτηση προς την Επιτροπή για το ίδιο ακριβώς θέμα. Εδώ λοιπόν έχουμε σαν κύριο μέλημά μα τι μικρές και μεσέ επιχειρήσεις. Έχουμε ένα κοινό μέλημα. Και ένα από τα ερωτήματα που θέτουμε είναι τι πράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει και οικονομικά αποτελεσματικά μέτρα στο μέλλον ε, που θα ενισχύουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι το νομοθέτημα, το πρόγραμμα SIP, πρόγραμμα για την κοινοτομία. το κοινό στρατηγικό πρόγραμμα πλαίσιο. Πώς θα διαμορφωθεί τώρα, τι ευκαιρίες δηλαδή μέσα στο πλαίσιο αυτό μπορούν να έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να διευρυνθεί η έννοια της ε, καιροτομία τόσο ώστε να συμπεριλάβει κάθε δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει και να ε, ρηπέσουμε στο σφάλμα να υποστηρίξουμε μόνο τις μικρομεσαίες εκείνες επιχειρήσεις ε, ως ανταγωνιστικές οι οποίες παρουσιάζουν άκρος ιδιαίτερη ε, καινοτομία, άκρος ξεχωριστή δηλαδή καινοτομία. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω να ληφθούν σωστά σταθμισμένες, ορθές αποφάσεις για το θέμα αυτό και κυρίως με, ε, σε σχέση με το ποιο κριτήριο θα χρησιμοποιηθεί και πώς μπορεί να ενισχυθεί η απλούστευση και η κατάρριξη γραφειοκρατίας. Το ΣΥΠ είναι λιγότερο γραφειοκρατικό γραφειοκρατικά ευερημένο από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και πιστεύω ότι ε, δεν ε, θα πρέπει να επιδεινώσουμε τις συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ας βρούμε λοιπόν έναν τρόπο πρακτικό, ας βρούμε μια λύση για το καλύτερο, για το βέλτιστο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να συνεχιστεί το πρόγραμμα ΣΥΠ και ώστε να μην καταλήξει τελικά να αποτύχει μέσα σε μια διαδικασία επανοργάνωση. Ευχαριστώ κύριε Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους μου για τη συμβολή τους σε αυτό το πολύ χρήσιμο ψήφισμα και να δηλώσω ότι συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες για ένα-δυο ζητήματα που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να είναι επικοδομητικές και χρήσιμες συμβολές για το τελικό κείμενο. Καταρχήν, στο κείμενο δεν αναφέρεται στις, επιπτώσει τη επιπτώσεις της παράνομης ε, εμπορίας από πλευράς των μικρών επιχειρήσεων. Δυστυχώς το λαθεμπόριο είναι κάτι το οποίο συχνά γίνεται από τις μικρές επιχειρήσεις και είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξη και των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων. Δεύτερη μου παρατήρηση αφορά τη την δεύτερη ευκαιρία και τη σχετική πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο οικονομικών δυσχεριών είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ και να βοηθηθούν να αναπτυχθούν. Αυτό με οδηγεί στην τελευταία μου παρατήρηση ε, νομίζω πως είναι λυπηρό που λίγες, κάποιες μάλλον από τις κοινοτόμες μας επιχειρήσεις που ήταν ΜΜΕ έχουν εξελιχθεί σε μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις πλέον και υπάρχουν πολύ λιγότερος ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη από ό,τι στις ΕΠΑ. Σημαντική ανάπτυξη αυτών των ΜΜΕ παρεμποδίζουν αυτές τις ίδιες να υιοθετήσουν καινοτόμα μοντέλα ε, επιχειρηματικά και νέες τεχνολογίες. Και γι' αυτό θα πρέπει να ε, καλλιεργήσουμε το πιο ρηψοκίνδυνο πνεύμα που υπάρχει στη ΣΥΠΑ και στη νέα γενιά των Αμερικανών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να το μεταφέρουμε εδώ εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς η κυρία Γιώρη, όπως ξέρουμε, έχει πάσχει από αφωνία και ο, ο υπάλληλος δεν επαστήβασε την απάντησή της. Elnök úr, biztos úr, tisztelt eh, képviselők! Κυρίε και κύριοι βουλευτέ. Θα ήθελα να κλείσω την ευγνωμοσύνη μου προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ενδιαφέρον του για την νομοθεσία τη σχετική με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και για την πρωτοβουλία αυτή να συζητήσει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ε, επί τη ευκαιρία της αναθεώρησης της σχετικής πράξης του Small Business Act δηλαδή, SBA. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα το οποίο στόχο έχει να ε, διαμορφώσει ένα πιο ευνοϊκό επιχειρησιακό περιβάλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία ε, των επιχειρήσεών μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν πολλούς εργαζομένους, εργαζομένους στην Ευρώπη, πάνω από 50 εκατομμύρια. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μέσω αυτής η πλήρης εφαρμογή του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις, του Small Business Act, αποτελούν προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία. Η επιτυχία της στρατηγικής μας για την ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες θα επηρεάσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ανάπτυξή μας άρα συναρτάται με τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει ε, καινοτόμου και ανταγωνιστικέ μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γι' αυτό καλωσορίζουμε την ε, ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ε, δημοσιεύθηκε το Φεβρουάριο του 2011. Στην ανακοίνωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέες πρωτοβουλίες για περαιτέρω δράση σε διάφορους ε, τομείς προτεραιότητας πρωτοβουλίες οι οποίες ακολουθούν ε, εκταμένες ε, διαβουλεύσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιες αρχές, των δημοσίων επιχειρήσεων και ως εκ τούτου ε, αποτελούν μια πιστή καταγραφή πιστεύουμε των προθέσεων και αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Συμβουλική και η Επιτροπή σε μια άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Ανταγωνιστικότητας στον Κούντελε της ε, Ουγγαρίας στις 13 Απριλίου συζητήσανε τα θέματα αυτά και ε, υποστήριξαν οι Υπουργοί, εξέφραν την υποστήριξη του Υπουργοί για τις προτάσεις της Ουγγρικής Προεδρίας. Ε, η προτεραιότητα λοιπόν που δίνεται είναι στην ΕΦΗ e e νομοθεσία Smart Regulation, χρηματοδότηση, ε, ε, διακυβέρνηση και ε, παγκοσμιοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να προβληθούν ως προτεραιότητες. Ωστόσο θέλω να επισημάνω ότι η Προεδρία πάνω απ' όλα ενδιαφέρεται να διατηρήσει την ορμή που έχουμε αναπτύξει με αυτήν την πρωτοβουλία και έτσι όταν έρθει η ώρα να συζητήσουμε στις 30-31 Μαΐου να λάβουμε αποφάσεις ουσιαστικές που θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε περαιτέρω. Στη συνεδρία σε αυτή τη 30-31 Νοεμβρίου πιστεύουμε ότι θα έχουμε δυνατότητα να υιοθετήσουμε προτάσεις που θα ε, προωθήσουν τις βασικές μας αρχές όπως το Think Small First, την αρχή ε, πρώτα απ' όλα να κοιτάς τη λύση σε, μικρό, σε μικρές διαστάσεις. Ε, πρόταση που έχει προέλθει καταρχάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα σχέδιο κανονισμού, ε, προς το Συμβούλιο, το, ε, κανονισμού του Συμβουλίου του 2008 Πρόταση η οποία είχε καταρχάς σαν στόχο ε, να διευκολύνει την μικρομεσαία επιχείρηση να αναπτύξει δραστηριότητε της μέσα σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό ταυτόχρονα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μείωση του κόστους και ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη. Στο Συμβούλιο εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες ε, για κάποιες πτυχές της προτάσεως. Και παρά τις προσπάθειες της Σουηδικής και Βελγικής Προεδρίας δεν ε, κατέστη δυνατή επίτευξη συνενετικής λύσης. Διαβεβαιώ πάντως τους ε, και τους βουλευτές ότι η Ουγγρική Προεδρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο να εξασφαλίσει πρόοδο Στη ιδιαίτερα καρφώδεις πλευρές αυτού του θέματος και ότι δεν θα πάψουμε τις προσπάθειές μας στην ε, ανέβρεση μια ενός καλού αποτελέσματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρέιν έχει το λόγο. President, uh, honorable members. Uh, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλές ερωτήσεις έχουν τεθεί. Και θα απαντήσω στην ερώτηση εξ νόμου του συναδέλφου Αντιπροέδρου Αντώνιο Ταγιάννη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιστοιχούν στο 99% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και δημιουργούν τη μεγαλύτερη προσθέμενη αξία καθώς και τα δύο τρίτα του τζίρου τη. Ε, ε, στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες χρειάζονται λιγότερη γραφειοκρατία, ευκολότερη πρόσβαση στην χρηματοδότηση, πράσινες αγορές και δεξιότητες που να αντιστοιχούν στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Αυτές είναι οι αρχές πίσω από την δική μας πολιτική περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως αντιπροσωπεύεται στο πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ευρώπη». Στο πλαίσιο των ερωτήσεών σας έχω ήδη κάνει κάποιες απαντήσεις ε, στην αναθεώρηση η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να εκτιμούν συστηματικά τον αντίκτυπο τη νομοθεσία του στι μικρομεσαίες επιχειρήσει χρησιμοποιώντα το τεστ για τις ΜΜΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν συνεργάζονται για τη μελέτη τη εφαρμογή του τεστ για τις ΜΜΕ στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κομισιόν θα χρησιμοποιήσει αυτό το τεστ ω βάση για το σχεδιασμό επιπλέον μέτρων για την υποστήριξη τη εφαρμογή και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών. Επίσης, ολοκληρώνουμε αυτή τη στιγμή μια μελέτη για τα προβλήματα όσον αφορά τις, ε, τη διαδικασία ε, χρεοκοπία στα κράτη-μέλη, ε, την δράση των ομήλων στα κράτη-μέλη. Στόχο έχουμε τα κράτη-μέλη να σχεδιάσουν τα κατάλληλα μέτρα για να εφαρμοστεί ε, η αρχή Think Small First στις διοικητικές τους υπηρεσίες. Αυτό θα καταστεί δυνατόν ιδιαίτερα ε, επεκτείνοντας την online διοίκηση καθώς και την ενιαία θηρίδα σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στην αναθεώρηση. Κατά δεύτερο λόγο, ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης θα εισαχθεί. Η Κομισιόν έχει καλέσει τα κράτη-μέλη να ορίσουν ε, έναν εκπρόσωπο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τον κύριο την κυρία ΜΜΕ για να ε, παρακολουθεί την εφαρμογή του Small Business Act στα κράτη-μέλη. Αυτό αυτή η διαδικασία θα συγκεντρώσει σε μια ομάδα αυτούς τους ε, κυρίους και κυρίες που θα συναντηθούν για πρώτη φορά στη Βουδαπέστη 24-25 Μαΐου τρέχοντος έτους. Η ΜΜΕ θα είναι η βασική δικαιούχη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την μείωση του διοικητικού φόρτου. Η Κομισιόν έχει υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο προτάσεις για την μείωση του διοικητικού κόστους πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά 30%, πάνω από 30% όταν εφαρμοστούν και βασιζόμαστε στο Κοινοβούλιο ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι προτάσεις μας θα υιοθετηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα. Ορισμένες προτάσεις θα ωφελήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως η αναθεώρηση της ε, τέταρτης οδηγίας λογιστικής, η οποία όταν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αναθεώρηση τις πρώτη ε, λογιστικές οδηγίες θα διευκολύνει τα κρατημέλη ώστε να εξαιρούν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από ορισμένε λογιστικές τους υποχρεώσεις. Τέταρτον, το, η πράξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, διευκολύνει τις ΜΜΕ ώστε να αναλάβουν, να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της πάρκιας ενέργειας και να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την περιβαλλοντική αγορά. Επίσης ενθαρρύνει την καινοτομία και αυτό θα εφαρμοστεί προσέχοντας ιδιαίτερα τις ΜΜΕ, προωθώντας ε, την δικτύωση, τις ε, νέες τεχνολογίες και την αποτελεσματική χρήση ή την, ε, την νέα χρήση των πόρων. Αυτά μέσα στο πλαίσιο του δικτύου Enterprise Europe. Τώρα, ως ναυαρχίδα στις πρωτοβουλίες μας, και στην ατζέντα που έχουμε υιοθετήσει, η Κομισιόν θα αξιολογήσει τις μελλοντικέ ε, δεξιότητες που χρειάζονται στις μικρές επιχειρήσεις σε μια πρώτη μελέτη εντοπισμού των μελλοντικών δεξιοτήτων αναγκών ε, σε δεξιότητες ε, έχουμε σχεδιάσει μια σχετική, διαδικασία, μια σχετική μελέτη ε, η οποία μόλις δημοσιεύθηκε και εντοπίζει τις δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προβούμε για να εντοπίσουμε τις μελλοντικές δεξιότητες και να τις προωθήσουμε πιο αποτελεσματικά καθώς και να τις συμπεριλάβουμε πιο συστηματικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα για τις μικροεπιχειρήσεις και τις βιοτεχνίες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Πίτρο Πελή, ο Πρόεδρος. Και τώρα τον λόγο η κυρία Τελκαστηγιό Μπέρα. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε αυτό το κοινό ψήφισμα που αφορά την επανεξέταση της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ. Μια πρωτοβουλία που ανάγεται στον Φεβρουάριο και προέρχεται από την Κομισιόν. Θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλούς ορισμούς το τι πάει να πει ΜΜΕ αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το μέσο ε, συνάρθρωσης της ε, οικονομίας και στη περίπτωση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, αν αυτό, αυτός ο σύνδεσμος που είναι η ΜΜΕ τα πάει καλά, είναι ισχυρό, τότε πάει καλά η οικονομία, ιδάλω όχι. Επομένω, ε, γι' αυτό λέμε ότι οι ΜΜΕ γεννούν ευημερία για την κοινωνία. Να σα πω τρία θέματα τα οποία μου φαίνεται ότι είναι βασικά για να μπορέσει να πάει καλά αυτή η υπόθεση. Πρώτα-πρώτα, ε, αυτό το δίκτυο επιχειρήσεων να είναι ισχυρό επίση, να αγκαλιάσουν οι ΜΜΕ πληροφορική, καινοτομία, διακυβέρνηση ηλεκτρονική. Ε, αυτό το σύννεφο της πληροφορικής, το cloud computing που λέγεται, οπότε θα πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να γίνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις. Επίσης είναι πάρα πολύ βασική και η καινοτομία και για τις ΜΜΕ, ε, για το startup, για την εκκίνηση των επιχειρήσεων θα πρέπει να υπάρξουν κινήτρα και κατά τρίτο λόγο να προσέξουμε το ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να ε, έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν στην εσωτερική αγορά και όσον αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς και όσον αφορά το, το μεθοριακό εμπόριο, τα πάντα που αφορούν την εσωτερική αγορά σαν, σαν όφελος. Έτσι, να βοηθούνται και να έχουν ανταγωνιστικότητα. Τελευταίο δε, προσοχή. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεται το, η αξία, η προσθέμενη αξία του επιχειρήν. Να, γιατί δεν θα πρέπει να είναι αδύναμο το δίκτυο των επιχειρήσεων. Προσοχή επομένω να μπορούμε όλα αυτά να τα προωθήσουμε και θα τα πετύχουμε μέσα από το εξή την εκπαίδευση. Επόμενη κυρία Ρία Μαντουρέλη, ζητεί το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαντουρέλη. Ναι, όντω ε, αυτέ οι ΜΜΕ έχουν ένα πλεονέκτημα, Έχουν την ευελιξία ε, είναι ευκίνητε είναι πιο κοντά στον πελάτη και έτσι μπορούν να λάβουν αποφάσει πολύ γρηγορότερα. Πρόκειται για κάποιες ε, αρετές πάρα πολύ σημαντικέ σε μια σημερινή τέτοια συγκυρία κρίση, όπου είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να αποφασίσει, να ανταποκριθεί, να αποκριθεί γρήγορα και γι' αυτό και λέμε ότι είναι πάνω από το 90% των επιχειρήσεών μα στην Ευρώπη η ΜΜΕ. Είναι επομένω ένα πρότυπο αυτό το οποίο είναι χρήσιμο, ωραίο να το κρατήσουμε για ε, να μην έχουμε τις μετακαταστάσεις γιατί το να κλείσει να φύγει μια επιχείρηση αυτό έχει τραγικά αποτελέσματα για την απασχόληση. αυτό οπότε προσοχή γιατί θα πρέπει να μην έχουμε τροχοπέδες στις ΜΜΕ από πλευράς του κράτους. Οπότε γι' αυτό και σας λέω ότι τι πρωτοβουλίες αν την συζητούμε είναι πάρα πολύ βασικές για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν όλα αυτά τα μέτρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι ΜΜΕ στην Ευρώπη χρειάζονται κατεπηγόντως την απαραίτητη πολιτική βούληση. Αυτή μας οδήγησε στο ΜΜΕ. Χρειάζονται μέτρα ρεαλιστικά, μέτρα ουσιαστικά και όσον αφορά τους, τους δημόσιους διαγωνισμούς. Και χρειάζεται να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, ενημέρωση μέσω άρτιας πληροφορικής, μέσω των κατάλληλων website, όμως αυτά δεν φτάνουν. Θα πρέπει εμείς εδώ από τη θέση μας να βοηθήσουμε ούτω ώστε να, του, να βοηθούν από το κράτος, από το κράτος ε, να είναι κατά κάποιο τρόπο κάτι σαν θετική διάκριση υπέρ τους. Να αρθούν όλα τα εμπόδια που εμποδίζουν τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρος, και τρώει το λόγο ο κύριος Κρόιτσμαν. Κύριε Επίτροπε. Κύριε Πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο ότι πολλά ακόμα έχουμε να κάνουμε για να προχωρήσει η Ευρώπη στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίω και σε εθνικό επίπεδο. Χαίρομαι όμως που στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο Small Business Act και να ενοποιήσουμε τις επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι μπορούμε πιστεύω να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να ε, προχωρήσουμε με την ε, αναθεώρηση την οποία θα πρέπει σε δύο χρόνια μέσα να έχουν ε, θέσει εφαρμογή τα κράτη-μέλη. Αυτή η περίοδος στα κράτη τα οποία δεν υπάρχουν ιδιαίτερε δυσκολίε θα ήταν σκόπιμο να περικοπεί. Αντί για δύο χρόνια καθυστέρηση να πούμε ότι θα πρέπει να την ενσωματώσουμε σε ένα χρόνο. Το καθεστώ ιδιωτική εταιρεία. μέχρι στιγμή δεν έχει εξασφαλίσει συμφωνία και γι' αυτό ε, χαίρομαι για την ε, παρακολούθηση του θέματος από την Ουγγρική Προεδρία, η οποία φαίνεται να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία. Με τέτοια μεταρρύθμιση θα βοηθήσει ιδιαίτερα τις μεσαίες επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν πόρους και για τη θέσπιση τους, ε, για την ανακήρυξη του, καταστό, του καθεστώτος, ε, για την εξασφάλιση νομικών συμβουλών. Χαίρομαι, όπως είπα, για τη σημασία που αποδίδει στο θέμα η Ουγγρική Προεδρία. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να βοηθήσουμε και στη διαδικα... στις διαδικασίες για τις δημόσιες προμήθειες, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν τις απαλλάξουμε από τη γραφειοκρατία. Αυτό, αυτό είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στη συμμετοχή του σε δημόσιους διαγωνισμούς, σε δημόσιες προκήρυξεις. Πρέπει λοιπόν να εξαλείψουμε αυτή τη γραφειοκρατία και με την ευκαιρία αυτή να στραφούμε και στη χρήση των σύγχρονων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή των μέσων επικοινωνία δηλαδή του ίντερνετ. Ευχαριστώ. Κύριε Σπίνμπορν, ένα λεπτό. Το ο νόμο περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακριβώ αυτό στο οποίο θα έπρεπε οι πολιτικοί και οι νομοθέτε να εστιάσουν την προσοχή του καθώ προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τι οικονομίε μα. Οι ΜΜΕ στη δική μου περιφέρεια τη Ουαλία αποτελούν το 98% των επιχειρήσεων και είναι λιγότερο βέβαιε όμω, και οι δικοί μου ψηφοφόροι ελπίζουν ότι θα μπορέσουν να απασχοληθούν από αυτέ τι επιχειρήσει. Γι' αυτό και υποστηρίζω του φιλόδοξου στόχου για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και είμαι υπέρ αυτού του, της δοκιμής για τις ΜΜΕ για κάθε είδος νομοθεσία σε συνδυασμό με τα όσα κάνει η κυβέρνησή μας ε, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Όμως είναι σκόπιμο να είμαστε πιο φιλόδοξοι και να επιτύχουμε περισσότερα. Έχω δει μεγάλη δημιουργικότητα στην ε, Ουαλία. Αποτελεί ένα κόμβο για την πρόθεση νέων δραστηριοτήτων σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και στη δημιουργία κέντρων αριστεία και γι' αυτό και διερωτώμε για το πώς θα μπορέσουμε να ενθαρρύνουμε αυτές τις εξελίξεις. Μεγάλα προγράμματα όπως ε, το διπλώματα ευρεσιτεχνίας και η ψηφιακή ατζέντα θα προωθήσουν τις ΜΜΕ και θα δώσουν δουλειές στο λαό της Ουαλίας και ολόκληρης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κλάρκ. Εδώ αναθεωρούμε 10 αρχές για την ενιαία αγορά, αλλά βλέπουμε ότι η Βροζώνη καταραίει. Πώς μπορούμε να δώσουμε λοιπόν περισσότερες ευκαιρίες. Επίσης θέλει η ΜΜΕ να ωφεληθούν από τις αγορές τις ε, ανοιχτές. Μα ποιες αγορές. Εγώ ρώτησα τον κύριο Πίτροπο Άντρο ποια μέτρα θα εισάγετε για να βοηθήσετε τις ΜΜΕ και ε, όταν μίλησε στην Επιτροπή ε, μίλ δεν πήρα καμιά απάντηση, αλλά τώρα φαίνεται να έχω κάποιες. Η αναθεώρηση ακολουθεί πέντε κατευθύντε γραμμέ για τη μείωση της πίεσης ε, και του φόρτου στις ΜΜΕ. Αυτά είναι απλά η χρήση κάποιων υφιστάμενων νομοθεσιών. Θα έπρεπε να προταθούν νέοι κανόνες όπως ε, για τις ευρωπαϊκές ιδιωτικές εταιρείες και τις κρατικές ενισχύσει, Αυτό σημαίνει ότι τελικά ε, εξαρθρώνονται διάφορες νομοθεσίες. Εξάλλου, ο, Επίτροπος, ε, ο πρόεδρος της Επιτροπής το εδώ ότι η γραφειοκρατία στην ουσία στραγγαλίζει τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Κύριος Σφιεύκα, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι. Εδώ έχουμε περίπλοκη νομοθεσία. Αυστηρή. Δεν είναι ευέλικτη. Εγώ έχω δουλέψει πάνω σε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και θα πρέπει να σα πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια το να ε, διαιρούνται οι κείμενε διατάξεις ε, όσον αφορά ε, την αξιολόγηση την αξιολόγηση μιας κατάσταση πριν και μετά θεσπιστεί κάτι και να βλέπουμε πώ είναι δυνατόν να διευκολύνουμε αυτόν τον κλάδο τον κλάδο τόσο ζωτικό γι' αυτό το κάνουμε και πριν και μετά εφαρμοστεί μια νομοθεσία Επομένω, είναι πολύ σημαντικό αυτό για την οικονομία ε, είπαμε ότι το, μικρό είναι ευέλικτο και θα πρέπει επομένω να μπορέσουμε το κοινοτικό δίκαιο να το μεταφέρουμε στο ιστορικό δίκαιο των κρατών μελών και επίσης θα πρέπει για την γραφειοκρατία που βαραίνεται τι α, ΜΜΕ να το ελαφρώσουμε. Επομένως, ε, είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση αυτής της πρωτοβουλίας και έχει τονιστεί ότι πάρα πολύ συχνά το, το, το, γραφειοκρατικό βάρος είναι υπερβολικό. Έχουμε και ένα σωρό εποπτικές διαδικασίες οι οποίες εμποδίζουν τις ΜΜΕ να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους βεβαίω μπορούν και δημιουργούν νέε θέσει εργασία. Επομένω, είναι θεμητό το να αναρωτιέται κανεί, ετήρησε τα υπεσχημένα η Κομισιόν όσον αφορά τη γραφειοκρατία και τη μείωσή τη. Λέγαμε για μείωση κατά 25%. Επίση, συμφωνούμε ότι αυτέ οι διατάξει για την αναθεώρηση τη κειμένη νομοθεσία θα πρέπει να τύχουν θετική υποδοχή και από τα κρατημέρια και από την Κομισιόν. Διότι θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να έχουμε όλε αυτέ τι τροχοπέδε. Ελπίζουμε ότι θα αποκομίσουμε θετικά αποτελέσματα όταν εφαρμοστεί αυτό το νομοθέτημα. Επίση, θα πρέπει να τονίσουμε το πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο πετύχαμε από το Ευρωπαϊκό Ενοχικό Δίκαιο και επομένω χρειάζεται να υπάρξει εύστοχη δόκιμη νομοθεσία και όλα αυτά να μας οδηγήσουν και σε καινοτομία που την οποία να την απολαύσουν και οι ΜΜΕ και ευχαριστούμε πάρα πολύ ο πρόεδρος και το έντολο στην κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ξέρετε, το 2011 πήγαμε στο 9,5% ανεργία στην Ένωση και 8% στην Ευρωζώνη. Δηλαδή, για τους νέους επίσης σε σχέση με το σύνολο του, του πληθυσμού είναι διπλάσια η ανεργία. Επομένως, θα πρέπει να δούμε το πώς θα ενθαρρύνουμε τις ΜΜΕ, πώς το επιχειρηματικό πνεύμα θα το ενθαρρύνουμε. Χρειάζονται αυτοί οι επιχειρηματίες ένα κλίμα, ένα περιβάλλον ευμενές. Επίσης θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση σε μια συγκυρία κρίσης χτυπιούνται ΜΜΕ από το πόσο καθυστερούν χρηματοδοτήσεις. Και επομένως χωρίς καινοτομία δεν μπορούν να προχωρήσουν. Κατά 33% Επίση, συμμετέχουν στι δημόσιε συμβάσει η ΜΜΕ και σκεφτείτε πόσο σημαντικέ είναι αυτές οι συμβάσεις για το το Ευρωπαϊκό. Επομένω βλέπετε ότι θα πρέπει να στηρίξουν περισσότερε ΜΜΕ όσον αφορά τι δημόσιε συμβάσει. Και γι' αυτό θα πρέπει και η Κομισιόν και τα κράτη να κάνουν ό,τι χρειάζεται, τόσο ώστε μέχρι το 2015 τουλάχιστον το 50% των δημοσίων συμβάσεων να ανατίθενται ηλεκτρονικά ε, στις ΜΜΕ όπως προβλέπεται από την ομοθεσία που θεσπίστηκε το 2005. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ακόμα αυτά που έχουμε θεσπίσει δεν ε, εφαρμόζονται ε, και το 2008 είχε εξαγγείλει το πρόγραμμά της η Κομισιόν όσον αφορά ε, την ΕΤΕ. Η ΕΤΕ υποτίθεται θα χρηματοδοτούσε κατά 30 δις της ΜΜΕ. Αλλά και ένα δισεκατομμύριο ε, δάνεια θα έδιναν τα κρατημέλη της ΜΜΕ. Για πέστε μας Κομισιόν, σε ποια φάση βρισκόμεθα όσον αφορά την υλοποίηση αυτών των υποσχέσεων, γίνεται αυτή η χρηματοδότηση και γίνεται με τρόπο δίκαιο. Τρία εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης χάθηκαν παρά τις επενδύσεις ε, στην πολιτική στήριξη. Αυτό είναι ο απολογισμός πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας και της στρατηγικής 2020 στην οποία υποτίθεται Πρέπει να δοθεί στήριξη για το επόμενο πολίτες πρόγραμμα πλαίσιο 2014 με 2020. Οι Ευρωπαίοι πολίτες ρωτώνται σε τι χρησιμεύει η Ευρώπη αν δεν μπορεί να λύσει τα οικονομικά προβλήματα της Επίρου και δεν μπορεί να μιλήσει με μια φωνή για την εξωτερική πολιτική ούτε και για τα χρήματα. Εύχομαι ότι τα όσα μας είπε ο Επίτροπος Ταγιάννη θα υλοποιηθούν και ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να απλοποιήσουμε τη γραφειοκρατία, να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην πίστοση και να διευκολύνουμε τις διαδικασίες. Έχουμε φτιάξει, φτάσει σε μια συμφωνία σημαντική ε, μέσω της πολιτικής βούλησης. Σας στη διάρκεια της επόμενης, ε, μάλλον αν τελικά όλα αυτά είναι μόνο σε Καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τους μικρούς επιχειρηματίες που στην περιοχή μου, το Βένετο, ε, αυτοκτόνησαν για να μην δουν τη χρεοκοπία των επιχειρήσεών τους. Πολλοί από το Βένετο βρίσκονται εδώ επισκέπτε. Κυρία Κάρενς. Συγγνώμη, ο κύριος Κάρενς, το συγγνώμη. Δεν πειράζει, Πρόεδρε. Πολύ συχνά οι οικογένειες αντιδρούν κατά έναν τρόπο παράδοξο. Οι γονείς δηλαδή δίνουν πιο πολύ προσοχή στο παιδί που κάνει πιο πολύ πασαρία, που κλαίει πιο πολύ. Ε, αυτό συμβαίνει και εδώ, στον πολιτικό βίο. Τείνουμε να δίνουμε πολύ πιο περισσότερη προσοχή στις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν πιο πολλά λεφτά, που φωνάζουν πιο δυνατά, που μας λένε «Α, εμάς να κοιτάξτε». Ενώ θα έπρεπε να φροντίζουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις πιο ήσυχες. Mm-hmm. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι σαν μεγάλα δέντρα στην Ευρώπη. Δέντρα που όμως δεν φτιάχνουν δάσος. Ξέρετε ότι έχουμε τα τρία τέταρτα του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού στι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μερίδιο του ευρωπαϊκού ΑΕΠ προέρχεται από μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μεταστρέψουμε την προσοχή μα, να σταματήσουμε να ε, ακούμε μόνο τι μεγάλε επιχειρήσει που φωνάζουν δυνατά και να κοιτάξουμε τι μικρομεσαίες, αυτέ που έχουν πιο χαμηλή φωνή, αλλά απασχολούν του πιο πολλού εργαζομένους. Και παρακαλώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις υποσχέσεις που έχει δώσει για περικοπή του γραφειοκρατικού φόρτου υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι κάτι που μπορείτε να κάνετε κατά την αναθεώρηση τη νομοθεσία που υφίσταται ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βάλτσιτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το 2008 η πρωτοβουλία της ΜΜΕ γεννήθηκε. Βοήθησε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη ΜΜΕ στην Ευρώπη. Κάναμε βήματα προς τα μπρος. Μειώσαμε τη γραφειοκρατική τροχοπέδη Είχαμε και εκείνη την οδηγία για την υπερημερία. Σήμερα διαπιστώνουμε ότι Όμω δεν ανταποκριθινόμαστε ή στις προσδοκίε των ΜΜΕ. Χρηματοδότηση χρειάζεται. Βελτίωση της επιχειρηματικής, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δεν τα καταφέραμε αυτά πλήρω. Βεβαίω, το δίκαιο του καταναλωτή διαφέρει από χώρα σε χώρα. Και επομένω αυτό δεν βοηθάει. Ούτε μπορεί η κάθε εταιρεία να μεταφέρει τι δραστηριότητά και σε μια άλλη χώρα. Να, τι θα πει θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Έχουμε πτωχεύσεις πολλές και δεν έχουμε καταφέρει μας να βοηθήσουμε αρκετά παρά τις προσπάθειές μας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε να είναι ευκολότερη χρηματοδότηση. Και έχει φανεί ότι οι τράπεζες αντί να χορηγούν δάνεια τα καθιστούν δυσκολότερα στο να χορηγηθούν. Ούτε τα στοιχεία που χρειάζονται δεν έχουν οι τράπεζες που χορηγούν τα δάνεια. Επομένως, θεωρούμε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί καλύτερα τις εξελίξεις και να επανεξετάζει όπως τώρα την πρωτοβουλία της ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο, πιο αποτελεσματικό, πιο δόκιμο περιβάλλον για τις ΜΜΕ. Πρόεδρος. Έχετε διαδικαστικό, τι θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με το πρόγραμμα Εράσμος για τους νέους επιχειρηματίες, γιατί ελέγχθη ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή τους στην κρίση και μόλις άκουσα ότι η Κομισιόν θέλει να περικόψει την χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος. Μήπως θα είχε νόημα ακριβώς λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν μια μεγαλύτερη δυνατότητα για να μάθουν νέες τεχνικές του επιχειρήν. Ευχαριστώ. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο λοιπόν του, του μέλλοντος, προτεραιοτήτων του μέλλοντος, πώς θα μπορέσουμε να αναδιαδρώσουμε την κοινωνία μας και ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα βήματα, όχι μόνο σε σχέση με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, αλλά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και το πρόγραμμα εργασμού για του επιχειρηματίε που αναφέρατε είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα πρέπει να καταβάλουν ακόμα περισσότερε προσπάθειε για να διατηρήσουν τα προγράμματα αυτά και στο μέλλον να έχουμε καλύτερα εκπαιδευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες στον τομέα των επιχειρήσεων που θα μπορέσουν να εφαρμόσουν όλες τις θεωρητικές ιδέες τις οποίες εμείς εκφράζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην πράξη. Πιστεύω ότι η περικοπή τέτοιων προγραμμάτων δεν θα πρέπει να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βούτσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την μεταρρύθμιση του Small Business Act θα πρέπει να περιστρέφονται γύρω από τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος για τις μικρές και τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν και πέραν των συνόρων της χώρας τους. Σύμφωνα με την ανάλυση της Κομισιόν, σε πάνω από 50% των κρατών μελών είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να δημιουργήσει μια επιχείρηση σε τρεις μέρες όπως είχε διακηρυχθεί. Πολλά κράτη επίσης δεν έχουν καμία αξιολόγηση σε σχέση με τον αντίκτυπο της νομοθεσίας. Δεν εφαρμόζεται ο κανόνας επίσης του ενιαίου ε, χώρου, του, της ενιαίας υπηρεσία που ασχολείται με την αδειοδότηση. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εμπλέκεται περισσότερο στην ε, θα πρέπει να εμπλακεί περισσότερο στην εφαρμογή αυτών των ρητρών και οι μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου και σε κεφάλαια επιχειρηματική σύμπραξη και η έννοια του ενιαίου σημείου αναφορά σε κάθε κατοσμένο θα πρέπει να εξασφαλίσει την απλοποίηση των διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών. Για να μπορέσουμε λοιπόν να επιτύχουμε το στόχο του 75% αποσχολησιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020, είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε είναι ω γνωστό <clears throat> αυτέ οι οποίε τώρα απομίζονται πολύ μεγάλο πρόσθετο κόστο λόγω τη κρίση. Λοιπόν, μπαίνουμε στην διαδικασία Catch the Eye, οφθαλμοθυρευτική και φυσικά έχουμε ε, να αντιμετωπίσουμε και τους περιορισμούς χρόνου. Πρώτη είναι η κυρία Μπασέσκου Uh, Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους από όλες τις πολιτικές ομάδες και η κυρία Μπασέσκου είναι η πρώτη που έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. για να ε, απλοποιήσουμε και να ευκαμπτοποιήσουμε την ε, νομοθεσία για να λάβει υπόψη τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να εγγραφούν όλα αυτά τα εγχειρήματα στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020. Θα πρέπει να κάνουμε δυνατό με ένα ταχύ και ολοκληρωτικό τρόπο να λαμβάνονται υπόψη όλες αυτές οι δράσεις, για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μικρή κλίμακα. Θα πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή και στην χρηματοδότηση επίσης ε, σε μεγαλύτερη κλίμακα επιχειρήσεων που είναι ιδιαίτερα ενεργέ στον τομέα τη καινοτομία. Η Ρουμανία είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα εφαρμογή βελτίστων πρακτικών ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε το επιχειρήν. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται λέγεται Startup Business και το οποίο είναι χρηματοδοτημένο με 2 εκατομμύρια ευρώ και έχει σαν αντικειμενικό σκοπό να αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες και δυνατότητες μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων. Επίσης έχουμε ένα πρόγραμμα για την εφαρμογή τη αρχή να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση τη μικρομεσαίας επιχειρήση. Η κυβέρνηση τη Ρουμανία υποστηρίζει πλήρω τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο έδαφο τη. Κ. Κούτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσεις αναθεώρησης της Small Business Act συμπεριλαμβάνουν χαιρετισμούς για τις προόδους λέει, που έχουν γίνει από την αρχή μέχρι σήμερα. Υπάρχουν όμως και ορισμένα προβλήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη χρηματοδότησή τους και τα χρέη τους. Όταν θα μεταφερθούν στην εθνική νομοθεσία οι οδηγίες αυτές, η οδηγία αυτή, θα ξεπεραστούν στην πράξη τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η ίδια η Ένωση και θα υπάρξει πρόβλημα ορατότητος και διαφάνειας. Επίσης πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις θα έχουν οι νέες αυτές προτάσεις γενικότερα στη ζωή των ΜΜΕ. Ευχαριστούμε ο κύριος Πάσκα. Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τότε που εγκρίθηκε η Small Business Act και γι' αυτό ήταν καλό να κάνει, που έκανε αυτή την αξιολόγηση φέτος η Κομισιόν. Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός συνεκτικού και συνεπούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος τελικά δεν ξέρω αν πέτυχαν όμως. Οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζήτησαν και νέα μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε σε περισσότερο βάθος πώς εφαρμόζονται στην εθνική νομοθεσία, πώς μεταφέρονται στην εθνική νομοθεσία οι κανόνες αυτή στη χώρα μου. Η εθνική νομοθεσία αντιστέκεται πολύ στις αλλαγές και συμπεριλαμβάνει ακόμη, εγκρίνει πολλούς τρόπους παρεμποδισμού της λειτουργίας των ΜΜΕ Πρέπει να γίνει κάτι για να τις βοηθήσουμε. Ευχαριστούμε κύριο Σόμπερμαγερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντική η διευκόλυνση που προκύπτει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την ε, Small Business Act. Εγώ επίσης ε, εκφράσω την ικανοποίησή μου για την υποχρέωση να πληρώνονται οι, δημόσιοι, οι λογαριασμοί του δημοσίου μέσα σε 30 μέρες. Είναι πολύ σημαντικό για την ταμιακή ροή για τις μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση και επίσης θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα και η, το σύνολο των ρυθμίσεων για τις διαμεθοριακές ε, ενέργειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να υπάρξουν θηγατρικές εταιρείες και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η προσπάθεια και στο μέλλον, γιατί η Ευρώπη θα, έχει να, θα πρέπει να έχει στο μέλλον και καλύτερες συνδέσεις με άλλους εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με την ε, μεταρρύθμιση της ε, Small Business Act. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει μεγαλύτερη προσοχή στα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει όλο αυτό το πακέτο να εφαρμοστεί πλήρω και σε εθνικό επίπεδο <clears throat> οι μικρομεσαίες επιχειρήσει αντιμετωπίζουν προβλήματα, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Για πάρα πολύ καιρό έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικέ δυσκολίε παρά το γεγονό ότι είναι οι πιο καινοτόμε. Έχουν πολλές φορές ένα τεράστιο βάρος ρυθμίσεων και κανόνων στις οποίες πρέπει που πρέπει να εκπληρούν. Νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο να υπάρχει και ένα καθεστώς ιδιωτικού δικαίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε κανόνες οι οποίοι θα έχουν ευφυή χαρακτήρα και νομίζω ότι η αρχή του Just Once, η αρχή δηλαδή του να υπάρχει μονάχα ένα σημείο αναφοράς για την αδειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να τηρηθεί και θα πρέπει να <clears throat> κάνουμε τις απαραίτητες διαρρυθμίσεις σε τεχνικό επίπεδο για να μπορέσει να αλλάξει το επιχειρηματικό κλίμα. Κύριος Στέρι. Πράγματι, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση δεν θα δημιουργήσει οπωσδήποτε μια θέση εργασίας στην Ευρώπη. Όμως υπάρχουν ε, κάποιες ε, θέσεις εργασίας ε, εν μέρη λόγω ύφεση και εν μέρη λόγω γραφειοκρατίας οι οποίες παρακολύονται από τις μικρομεσαίες επιχειρώσεις. Χαίρομαι που σας ανακοινώνω ότι η κυβέρνησή μας ανακοίνωσε μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι που χαιρέτησε ο επιχειρηματικός κόσμος σήμερα θα υπάρχουν πιο ευφυείς ε, φόροι και δυνατότητες πρακτικής άσκησης, επί παραδείγματι. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε την απάτη, τι ε, οικονομία της μαύρης αγοράς ε, για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και επίσης θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα για ηλεκτρονικό εμπόριο και να υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πολλές νέες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τέλος, ο κύριος Σιλβέστρης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αναθεώρηση του Small Business Act αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία εάν ξεκινήσουμε από την προϋπόθεση ότι κατανοούμε πόσο πολύτιμο είναι όλο αυτό το κεφάλαιο το οποίο εκπροσωπούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο νότο της Ιταλίας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ικανή και αναγκαία συνθήκη για το παραγωγικό μέσο. Ε, στην περιοχή μου οι κλωστοϊφαντουργίες είναι ως επιτοπλίστων μικρές και μεσές επιχειρήσεις ε, τεράστιες ε, περιοχές της Υπέθρου τα περασμένα χρόνια ζούσαν χάρη σε αυτές τις μικρές και μεσές επιχειρήσεις. Σήμερα αυτές οι μικρομεσές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ακριβώς και λόγω του ανταγωνισμού και το γνωρίζουν και οι φοιτητές του Μπαρέτα που είναι εδώ σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει λιγότερη γραφειοκρατία, λιγότερο άχθος, ε, λιγότερες καθυστερήσεις στις αποπληρωμές και να υπάρχει και η σταθερότητα τη οποία έχουν μεγάλη ανάγκη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Ρεν. President. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ πολύ διότι κάναμε μια ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Αυτό επισημάνθηκε από αρκετούς ευρωβουλευτές και συμφωνώ πολίτες ότι η ευημερία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι υψής της σημασίας για την ανάκτηση της ευρωπαϊκής ε, ανάπτυξης ε, και οικονομίας. Όταν πηγαίνουν καλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πηγαίνει καλά και η ευρωπαϊκή οικονομία. Σας διαβεβαιώ ότι η εφαρμογή του Think Small First και οι προτινόμενες δράσεις ε, στο Small Business Act αποτελούν βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και σας ευχαριστώ και για την υποστήριξή σας επί του θέματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στη στενότερη συνεργασία με όλους τους ε, σχετικούς ε, φορείς, ιδίω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και αποτελεσματική εφαρμογή του Small Business Act σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων τον Οκτώβριο θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για να ε, γνωστοποιήσουμε τις ε, πολιτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την ε, Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Διοργανώνουμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αποκοινούμε το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα η κυρία Γιώρη αλλά μας ενημέρωσαν ότι έχει χάσει τη φωνή της. Δεν θα μπορέσει να μιλήσει. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δράση εδώ και τώρα είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Όπως είπε και ένας από τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σέβομαι και συμμερίζομαι απόλυτα τις απόψεις τους. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ακούσαμε πολλές φορές, είναι ένας από τους κυριότερους δημιουργούς θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης είναι απαραίτητο να αναθεωρήσουμε τις ιδέες μας για το πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η Ουγγρική Προεδρία πιστεύει σε μια κοινωνία <clears throat> και μια οικονομία που βασίζεται στην εργασία σε αξιοπρεπές επίπεδο και θέλουμε εμείς να βασιστούμε για αυτό το εγχείρημα πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το οικονομικό περιβάλλον έχει αλλάξει εκ βάθρων από το 2008. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν της ε, Small Business Act είναι πράγματι απαραίτητη. Εμείς χαιρετίζουμε την ε, συνένεση που ανέφερε ο κύριος Κόφερ μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και χαιρόμαστε πολύ για τον μεγάλο αριθμό βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οι οποίοι εξήραν τις προσπάθειες της Ουγγρικής Προεδρίας. Πρόκειται πράγματι για μια προτεραιότητα για την Ουγγρική Προεδρία. Επιτρέψτε μου να σας ε, αναφέρω ορισμένα επιμέρους θέματα. <clears throat> Μετά από αυτά τα οποία άκουσα από εσά, με μεγάλη προσοχή παρακολούθησα αυτά που ελέγξαν, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας πω ότι επί των αρχών υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και η ατμομηχανή της ανάπτυξη και της απασχόλησης. Το να αυξήσουμε λοιπόν την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων είναι η πρώτη προτεραιότητα για το Συμβούλιο. Αυτό αντανακλάται και στο, στα συμπεράσματα που θα εγκριθούν από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, λέει, προσεχώς. Στο τέλος Μαΐου, δηλαδή, και στα συμπεράσματα αυτά είναι ανάγλυφο το γεγονός ότι κάποια από τα προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στον τομέα του Small Business Act πρέπει να επιληθούν, όπως είναι η καλύτερη πρόσβαση της πιστός, καλύτερη χρηματοδότηση, καλύτερη πρόσβαση σε αγορές είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε παγκόσμιες αγορές και επιπλέον η μείωση του διοικητικού φόρτου, διοικητικού άκτους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαιρετίζουμε το γεγονός <clears throat> η οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές η οποία έχει πλέον εγκριθεί από το Συμβούλιο παροτρύνει τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία του ταχύτερο δυνατό, κάτι το οποίο θα ανακουφίσει και θα βοηθήσει ιδιαίτερα την κατάσταση ευσότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Χαίρομαι επίσης για το γεγονός ότι το Συμβούλιο είναι πολύ κοντά σε μια τελική συμφωνία <clears throat> επί τη βάση των στόχων που έχει θεσπίσει η Κομισιόν για τη μείωση του διοικητικού φόρτου επί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες αυτές, οι μικρομεσαίες εταιρείες θα μπορούν να δημιουργούνται μέσα σε τρει μέρε, να εγγράφονται στα Μητρώα μέσα σε τρεις μέρες με ένα κόστο χαμηλότερο από 100 ευρώ. Πάνω από 23 κάτι μέλη έχουν συνταχθεί με αυτή τη διαδικασία ενισχυμένη συνεργασία και αυτό θα μπορεί και προωθείται και η εξέταση του κανονισμού για τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο. Αυτό, αν πραγματικά καρποφορήσει, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Ο κύριος Κρόιτσμαν έθεσε και το θέμα της ευρωπαϊκής εταιρείας, του ευρωπαϊκού Καθεστώτο για τι εταιρείε. Εμεί θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί να Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο σε αυτό το θέμα και μονάχα μια δράξη κρατών μελών δεν έχουν ακόμα αποδεχθεί την ευρεία συνένεση που υπάρχει στο Συμβούλιο. Το να γίνει δεκτό αυτό το νομοθέτημα από όλου, αυτό θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπή για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στην Ευρώπη και η ελπίδα μα είναι ότι θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να προχωρήσουμε και ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ασκήσει και πίεση στα υπολοιπόμενα κράτη-μέλη για να μπορέσει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εμείς έχουμε συζητήσει ήδη με τα μέλη τη Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων που είναι η φυσική μα σύμμαχη για αυτό το θέμα. Α πω τώρα κάτι και για τη στρατηγική του 2020. Ο στόχος, η στόχη καλύτερα, που περιλαμβάνεται στη στρατηγική <clears throat> της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα μέτρα και να υλοποιούνται σε συγκεκριμένα εγχειρήματα τα οποία θα βοηθήσουν την κατάσταση των μικρόμεσών επιχειρήσεων. Φυσικά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πράξουν τα υπεσχημένα, δεν αρκεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρξει και σε εθνικό επίπεδο μεγαλύτερη απλοποίηση και τα φορολογικά συστήματα θα πρέπει να γίνουν φιλικότερα προς, τα, προς τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Πολλά κράτη έχουν πράξει κάτι τέτοιο και κυρίως η Ουγγαρία που προεδρεύει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα τη συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 12. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο, στη δήλωση της Κομισιόν και του Συμβουλίου για την εξέλιξη της κρίσης χρέους